Good afternoon. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε ώστε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου. Οπότε περνάμε στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης 2019. Η συγγήτρια η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 Not all members are... Δεν ψήφισαν άλλοι. Είναι όλοι εντάξει, όχι. Είστε έτοιμοι υπέρ της ψηφοφορίας. Τέλεια. Ας προχωρήσουμε συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. εποχές, Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Close the vote. Πέρας Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά Close the vote. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. 28 in favor. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Close the vote. Πέρα ψηφοφορία. Δεν κρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. G. Κατά. Αποχέ. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήταν σαφές. Vote is open. Vote is closed. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφοφορίας. It's tight vote and it means it's rejected. That's... Απορρίπτεται από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου λένε, με αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε πάμε στην τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε 96 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ψηφοφορία. 28-27 εγκρίνεται Πάμε στην 72. it correct. Approve. Um, sorry. In favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται να εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. You can check them also, or you do them all electronically. Yes. The vote is open. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. And then now we... Πάμε στην 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 23-28, απορρίπτεται. 106. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. It's clear. No, it's... Είναι σαφές. Μου φάνηκε ότι απορρίπτεται. Ναι, ωραία, απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 ε, 188 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Open the vote. Close the vote. ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Σαφώς απορρίπτεται. 19.33. Πάμε τώρα στην 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 101. Να τις κάνουμε όλες ηλεκτρονικά για να είναι πιο εύκολο για να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για ποια? Για την 101. 101. Ζητά συγγνώμη ομιλήτρια. 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 107. Α, έρχεται η ψηφοφορία. Να περιμένουμε λίγο. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 85. Άρχιδη ψηφοφορία. Mm. ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H ή τα. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορια ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 169 από τις συμβαστικές άρχιδες ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική και άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική κάπα. Άρχεται, πέρας. Adopted. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 119. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική έλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική νη. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Τροπολογία 45. Υπέρ... Ε, άρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Compromise P. Συμβιβαστική P. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. συμβεστική S. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία τώρα. Να εξηγήσω γιατί στο αρχικό κείμενο είχαμε επενδύσεις άειλες και υλικές ε, και εγώ πρότεινα ότι αφού είμαστε στην ε, Επιτροπή Οικονομικών να πούμε επενδύσεις ε, που σχετίζονται με την μετάβαση ε, δεν έχει νόημα να πούμε άειλα και υλικά αντιρρήσεις ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία πρέπει να ψηφίσετε την τροπολογία με την προφορική και αν καταπέσει πρέπει να ψηφίσετε την αρχική συμβιβαστική. Εγώ έλεγα ότι είμαστε κατά, αλλά θέλουμε να ψηφιστεί. Όπως κάνουν οι σωστοί συνάδελφοι. Το εκτιμάμε. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε τη συμβιβαστική χωρίς την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται τροπολογία 193 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική U. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 2.28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 229. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 230. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.31 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 2.32 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 2.33 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 2.34. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.35. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.27 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται πάμε τώρα στην 2.49 άρχεται ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική W. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 248. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική χ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ύψιλον Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ζήτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζήτα, ζήτα, λέει ο πρόεδρος. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σα, κυρία Πρόεδρε. Μισό λεπτό δώστε μας, παρακαλώ, γιατί κάποιε τροπολογίε υιοθετήθηκαν κατά των συμβαστικών τροπολογιών και πρέπει να αξιολογήσω, αλλά μπορώ να το κάνω σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Λογικό μου φαίνεται. Καλώ. Παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Νομίζω ότι πέρασε το ένα λεπτό και δύο και τρία θα έλεγα. Παρακαλώ καθίστε λοιπόν. Για να προχωρήσουμε. Okay. Okay. Can we move on and vote on the text? Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 18 in favor, 34. 34 κατά 18 υπέρ, 4 αποχές. So, let me just remind you that we will meet Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι θα συνεδριάσουμε αύριο στις 9 για τις ακροάσεις, ε, για την ακρόαση του Πάολο Τζεντιλόνι. Ευχαριστώ όλους.